Σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση του σχεδίου. Ημερήσιας διάταξη υπάρχουν τροπολογίες, όχι. Μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Σημείο 2. Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. για το σημερινό θέμα τι, έχει, τι προβλέπετε ότι τα θύματα βίας έχουν δικαιώματα μεταξύ των οποίων είναι και η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Και Γι' αυτό είναι θέμα ε, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα και της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Αποφάσισαν λοιπόν οι δύο ε, επιτροπές να συνεργαστούν στενά και δυνάμει το άρθρο 51 να διοργανώσουν και μια κοινή συνεδρίαση. Κάνουμε λοιπόν αυτήν τη συνεδρίαση όπου προεδρεύουν και οι δύο πρόεδροι, δηλαδή ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και εγώ η ίδια από την Επιτροπή Γυναικών. Ε, πέντε κράτη-μέλη τον Ιανουάριο ανέλαβαν μια πρωτοβουλία ε, για ε, οδηγία η οποία υπευλήθη στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συγητές ε, στο Κοινοβούλιο έχουν ήδη υποβάλει τις εκθέσεις τους και οι βουλευτές έλαβαν γνώση της θέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Επίσης, ε, ε, λάβαμε και την γνωμοδότηση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σχετικά με τη νομική βάση της οδηγία. Στις 4 Ιουνίου συζητήθηκε στη κοινή συνεδρίαση η πρόταση οδηγία. Είχαμε στις 12 Ιουλίου την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 141 ε, τροπολογίες υπευλήθησαν και 12 συμβαστικέ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λόπες Αγγιλάρ που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών όπως σας έλεγα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Εάν όχι θα ακούσουμε τους δύο εισηγητές μας. Διαδικαστικό είναι. Ναι, θέλω να σας πενθυμίσω ότι υποτίθεται θα ψηφίζαμε ε, στις 9. Ε, πολλοί όμως θα έρθουν στις 10 από τη δική μας την Επιτροπή. Μπορείτε παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Όπως έλεγα, θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές μας. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ από την Επιτροπή Γυναικών. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ε, ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που θα ήθελα να κάνω να ευχαριστήσω πρωτίστως την άλλη εισηγήτρια, την κυρία Ρομέρο, με την οποία συνεργαστήκαμε. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδες ηγητές και την γραμματεία καθώς και τους βοηθούς που μας συνέδραμαν στο έργα μας. Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για τα θύματα γιατί κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος και ε, πιστεύω ότι με αυτό το κοινοβούλιο αποστέλουμε ένα ηχηρό μήνυμα συνδρομής προς τα θύματα, όχι μόνο τα θύματα της βίας, αλλά κάθε ε, μορφής ε, διάκρισης, όλες όσες μορφές που ανακλώνουν που εκφράζονται σε, αυτό, σε αυτή την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θερμό ευχαριστώ λοιπόν και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρομύρο από την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. <clears throat> Eh, Και εγώ επίσης θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές που μας βοήθησαν να βελτιώσουμε την έκθεση. Επίσης όλους όσους ε, μας ε, βοήθησαν ειδικά τον εισηγητή από το ΕΛΚ που συνέβαλε στην πρόθεση αυτής της πρωτοβουλίας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Σήμερα πράγματι όπως ε, τόνισε η Τερέζα Χιμένε Θεστερίλ, είναι πράγματι μια μεγάλη μέρα για τα θύματα και ελπίζουμε το μήνυμα αυτό όχι μόνο να φτάσει στα ίδια τα θύματα που είναι οι πρώτοι που θα ευεργετηθούν από αυτά τα μέτρα, αλλά να είναι ένα μήνυμα που θα εισακουστεί και από το Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει αυτά τα μέτρα. Η Βελική Προεδρία θα πρέπει να δώσει μια σημαντική όθηση προς τα μπρος και ελπίζουμε να εγκριθεί, να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια πριν από το πέρας της Βελγικής θητείας. Σας ευχαριστούμε και πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάνουμε μια ενδεικτική ψηφοφορία για να λάβουμε εντολή διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Είναι ψηφοφορία προς ανατολισμού, orientation vote στα αγγλικά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Start with compromise. Αρχίζουμε με τη συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συζητώ συγγνώμη, ε, ξέχασα, λέει η Πρόεδρος, την ε, συμβιβαστική τροπολογία υπεριθμών 5. Συμβιβαστική 5 λοιπόν, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 33. Α, εγκρίθηκε 33. 34. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές α καταπίπτει okay. Okay. We vote 142 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 Α, ναι, έλεγχος. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για την 147. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Μπορείτε να δείτε τώρα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην οθόνη. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπαρθμόν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει Άρα πάμε στην 166 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να κάνουμε μια επαλήθευση για την 167 ε, ψηφίστε παρακαλώ The ψηφοφορίας 42 υπέρ, γιατί είχαμε και την ψήφο του κυρίου Λόπες, λέει η Πρόεδρος, 30, ε, 30 μία ψήφη υπέρ εννοεί μάλλον, 34 κατά, απορρίπτεται. 46, 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 ε, υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ επαλήθευση ε, ψηφοφορία ...168, έτσι. Πέρας. 39 ψήφοι υπέρ 28 κατά και μία αποχή. Εγκρίθηκε λοιπόν. 48 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 καταπίπτει πάμε στην 170 υπέρ ένα λεπτάκι διορθώνει η πρόεδρος ένα λεπτό 148 on 170 uh, because 148 fell. Yes, so we go to So we go to 173. Yes. So we go to amendment. Τώρα πάμε στη τροπολογία 173. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 Α, καταπίπτει λέει πρόεδρος, λοιπόν. Και πάμε στην 178 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα φτάνουμε στη συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 223 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές Νομίζω πρέπει να γίνει επαλήθευση. Για την τροπολογία 223, 223 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 42 ψηφί υπέρ. Όχι, 43 υπέρ, 28 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. 57 ε, τμήμα 1. Σε τρία τμήματα είναι. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Α, καταπίπτει. Ναι, ναι, καταπίπτει. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190. Καταπίπτει. 191 Αποσύρεται μάλιστα. So we go to amendments. 194 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 196 ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Οι σοσιαλιστές έχουν, είναι υπεράριθμοι, έχουν μία ψήφο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Κάποιος από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ, δεν μπορεί να ψηφίσει. Α, τώρα ρυθμίστηκε, ρυθμίστηκε, πέρας ψηφοφορίας. 32 ψήφοι υπέρ. 33 διορθώνει ο Πρόεδρος. Και 37 κατά και καμία αποχή απερίφθη. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 198 υπέρ, κατά αποχές Απεορίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 61 τμήμα 2 τώρα ε, καταπίπτει 62 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 210 τμήμα τρίτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για τη 220 πέρας εγκρίνεται με 10 θες 39 πέρα 30 κατά εγκρίνεται ...79 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...80 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 228 υπέρ κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 228 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 35 υπέρ, 33 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. Ναι κυρία Γιανακουδάκη. Κάποιες τροπολογίες μου, η 219 την ξεχάσατε. Σίγουρα θα θέλετε να υποστηρίξετε και θέλω να σας δώσω αυτή τη δυνατότητα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, λέει η πρόεδρο. Πρώτα σε αυτό που είπε η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Λοιπόν, καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι υιοθετήσαμε, εγκρίναμε το σημείο για τις 20 ημέρες Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε την τροπολογία. Σε αποφασίσαμε για τις 20 ημέρες ήδη πριν τη 2.19. Ο κ. Σταραμπέλα. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, είναι τροπολογία 215 προβλέπει τις 20 ημέρες εγκρίθηκε, οπότε καταπίπτει η 2.19. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πάμε στην 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 κατά τμήματα, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά από Πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ ψηφίστε το δεύτερο τμήμα της 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 230 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 230. Ξεκινάει η ψηφοφορία μας. Τέλος ψηφοφορίας. 35 υπέρ, λέει πρόεδρος, 34 κατά εγκρίνεται. Έχει λήξει η ψηφοφορία και έχουμε αποτέλεσμα. Yes. Yes, Κυρία Λούλινγκ. Αν σηκώσετε το χέρι σας την επόμενη φορά που θα ψηφίζουμε θα μπορέσουμε να σας δούμε. Πριν έχετε στα χέρια σας την κάρτα. Η κυρία Λούλινγκ, το είπα από την αρχή. Να είστε δίκαιοι. Πέρα, τώρα ψηφίσουμε την τροπολογία 88, λέει η πρόεδρο. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ α καταπίπτει We go to amendments number two. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να διεξαχθεί έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 93. Κυρία Λούλινγκ, ναι. Τέλος ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 41 κατά, απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται έλεγχος για την συμβαστική 12 ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 65 με 5. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος όσον αφορά την τροπολογία 5. Ξεκινάει ο έλεγχος. Ψηφίζουμε. Τέλος. 41 ψήφοι υπέρ. 30 κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Ε, Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 104. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote is closed. Πέρας. 36 υπέρ, 35 εκατά. Υιοθετείτε. 106. 106. παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Κατά τμήματα. Τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχή ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία και αφορά την τροπολογία 10 The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 31 κατά, εγκρίνεται, 108 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο Η 10 εγκρίθηκε, οπότε καταπίπτει 109. Οπότε. Όχι, πάμε στην 109 μάλλον, λέει η πρόεδρο. Yes. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ, κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο όσον αφορά τη 15. Ξεκινάει ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα 40, 40 υπέρ, 30 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην αριθμό υπαριθμών 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές νομίζω πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την 111 ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος Πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 31 ψήφι κατά, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε, θα ελέγξουμε. Για την 113 ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει τώρα. Πέρας. 40 υπέρ, 31 κατά, οπότε εγκρίνεται. Και έχουμε συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 ηλεκτρονική ψηφοφορία θα δεξαχθεί τώρα όσον αφορά την τροποποιημένη πρόταση. Ξεκινάει η ψηφοφορία η ηλεκτρονική. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Θερμά συγχαρητήρια και στις δύο εισηγήτριες και στους δύο εισηγητές και συγχαρητήρια σε όλους μας γιατί υπάρχει περαιτέρω τώρα προστασία για τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Τώρα ε, θα συνεχίσουμε αλλά θα ήθελα εξ ονόματο τη Επιτροπής των Γυναικών να ευχαριστήσω και του εισηγητές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και όλους τους συναδέλφου και τη Γραμματεία από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την αγαστή μας συνεργασία για αυτό το θέμα κοινή αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Um, τώρα έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών που θα αρχίσει, οπότε αποχωρήστε όσοι είναι να αποχωρήσετε. we will start our committee meeting. Θα αρχίσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών.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 Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Γυναικών. Σημείο 3. Έγκριση της μερίσιας διάταξης. Ε, για το σημείο 12 θα αναβληθεί η συζήτησή του γιατί άλλαξε το χρονοδιάγραμμά της η αρμόδια επιτροπή. Άλλες αλλαγές δεν έχουν σημειωθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, οπότε το θεωρώ εγκεκριμένο. Ωραία, τέσσερα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διόρισε τη Μισελ Μπασελέτ, πρώην πρόεδρο της Χιλής, ε, για να ηγηθεί ε, της νέας υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις γυναίκες. Εξ ονόματος της Επιτροπής ε, θα αποστείλουμε συγχαρητήρια επιστολή στην νεοδιοριστήσα πρόεδρο της, του νέου, της νέας υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις γυναίκες. 5. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 14 Ιουλίου 2010. Εάν δεν ε, προκύψουν στάσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα εγκριθούν τα πρακτικά αυτόματα. Ε, σημείο 6. Ανακοινώσεις σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών ε, κατά την χτεσινή συνεδρίαση. Η ομάδα SD, οι σοσιαλιστές, θα εκδώσουν έκθεση σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση Επίσης, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Απασχόλησης σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής για την αγορά εργασίας και τα κοινωνικά πρότυπα. Θα υποβάλουμε τροπολογίες απευθείας στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Το ίδιο θα κάνουμε και για την κοινή διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την ε, έκθεση για την ανάλυση αντικτύπου ε, αποφάσισαν οι συντονιστές, η Πρόεδρος, να συντάξει μία επιστολή προς τον αρμόδιο για αυτήν την χνομοδότηση Αρχίσαμε να συζητάμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών για το 2011 και για τις επίσημες ακροάσεις αποφασίσαμε να γίνει ακρόαση για τις ε, γυναίκες μόνες, ε, για τις γυναίκες και τις κλιματικές αλλαγές, ε, για την Τουρκία και την ισότητα και για την κατάσταση των γυναικών, κατάσταση ένοπλης σύραξης ή πολέμου και για την ισότητα των δύο φύλων. Αποφασίσαμε για τις αποστολές που θα γίνουν το 2011 για τη Βαρσοβία παραδείγματο χάρη για να προετοιμάσουμε την Πολωνική Προεδρία και μία άλλη αντιπροσωπεία στην Κοπενχάγη εν ώψη της Δανικής Προεδρίας. Επίσης αποστολή προς την Κροατία και θα θέλαμε επίσης να κάνουμε μία, μία αποστολή στην Παλαιστίνη. Επίσης για το 2011 και την Παγκόσμια ημέρα γυναικών το θέμα θα είναι ο ρόλος των γυναικών στην μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση όπου συμπεριλαμβάνουμε και το ρόλο των γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν από την Πρόεδρο να συντάξει επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, αναλύσεις αντικτύπου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την, ε, γονική, για την άδεια μητρότητας. Θα ζητήσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα τονίσουμε ε, ότι ήταν ε, εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση να μην υπάρξει υπέρβαση του ε, χρονοδιαγράμματος, να, έχουμε, να λάβουμε γέρο στο σχέδιο, γιατί εμείς είχαμε προγραμματίσει τη συζήτηση για την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν για την συνάντηση, τη χθεσινή συνάντηση των συντονιστών. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 7, ο αντίκτυπος διαφήμισης συμπεριφορά των καταναλωτών. Το Μάρτιο του 2010 αποφάσισαν οι συντονιστές να εκδοθεί έκθεση ε, προς ε, την Επιτροπή ΤΡΕΙ για σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης συμπεριφορά των καταναλωτών και από την Επιτροπή μας ε, η συντάκτρια είναι η κυρία Παπαδοπούλου και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Παρακαλούμε κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους, ε, όλες τις σκιώδεις εισηγήτριες από όλες τις πολιτικές ομάδες και όλους τους συναδέλφους βουλευτές που με τις 40 περίπου τροπολογίες που εισηγήθηκαν έχουν βελτιώσει την παρούσα γνωμοδότηση, η οποία ακριβώς αφορά τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Είναι μια γνωμοδότηση η οποία επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς τα θετικά της σωστής διαφήμισης με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, στην προσωπικότητα της γυναίκας, χωρίς ε, σεξιστικές αναφορές και χωρίς στερεότυπα. Θεωρούμε ότι με τη συμβολή όλων ε, το κείμενο που έχουμε ενώπιον μας για γνωμοδότηση ε, είναι σαφώς ενισχυμένο και ευχαριστώ θερμά τον Γραμματέα της Επιτροπής όπως επίσης και τις κοινοβουλευτικές μου συνεργάτηδες που εργάστηκαν για αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Έχουν επιτευχθεί 8 συμβιβαστικέ τροπολογίες και ευελπιστώ με την ψήφων όλων των παρευρισκομένων ότι θα περάσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ να επαληθεύσουμε τη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 6 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Εννέα ψήφοι υπέρ, 11 ψήφοι κατά, συνεπώς απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 12 ψήφοι κατά και 9 ψήφοι υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές νομίζω θα πρέπει να επαληθεύσουμε 28 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 12 ψήφοι κατά και 9 ψήφοι υπέρ. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Συμβαστική 7. Άρχεται ψηφοφορία. Vote. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 11 ψήφοι κατά και 9 ψήφοι υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν. Και τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά να γίνει έλεγχος για τη 33 επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 11 ψήφοι υπέρ και 12 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Και τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία επαριθμό 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίν, ε, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 Συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε την ψηφοφορία για την παράγραφο 5, τροπολογία 35 της κυρία Σίλβια Κώστα. Μα γίνει επανάληψη. Ε, Είναι αυτή η ψηφοφορία που κάναμε. Αν έχετε την καλοσύνη να την επαναλάβετε παρακαλώ. Λυπούμε. Αλλά, κυρία Πατέρα, όταν έχουμε καταλήξεις, έχει γίνει ψηφοφορία, δεν μπορούμε να την ξανακάνουμε. Έχει λήξει η ψηφοφορία. Λυπούμε. Συγγνώμη. Έγινε περασμένη ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών όπου κάνατε μια επανάληψη ψηφοφορίας και είχα ζητήσει και είχε γίνει επανάληψη. Υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορούν να είναι μάρτυρες ότι έγινε αυτό. Ήταν στην προηγούμενη ψηφοφορία που είχε επαναληφθεί σε ένα σημείο. Δεν θυμάμαι λέει ο Πρόεδρος Υπάρχει τεχνικό, θα υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, τώρα πράγματα είναι ξεκάθαρα και πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία και ψηφίζουμε 37. Περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κυρία Ματήρα. Κοιτάξτε, είχα αφαιρεθεί για μισό λεπτό και κάνει την ψηφοφορία. Δεν ψήφισα ούτε σε αυτή την περίπτωση. Ε, Λοιπόν, ε, λοιπόν, αυτή τη φορά μπορούμε να επαναλάβουμε, διότι δεν πρόλαβα. Και δεν έχει εκφραστεί για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στην συγκεκριμένη ψηφοφορία. Αυτή μπορούμε να την επαναλάβουμε. Ε, μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 37. Άρχεται η ψηφοφορία για την 37. πέρας της ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. 10 κατά, 9 ψήφοι υπέρ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα τη 39 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να γίνει επαλήθευση, ναι, γιατί την 39 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 10 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά και 7 αποχές. Τώρα θα ψηφίσουμε τις 40 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει επαλήθευση για τη 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Να ξεκάθαρο αποτέλεσμα. 20 υπέρ, 3 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, ε, τροπολογία υπερθμών 1. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 ψήφισαν υπέρ, 3 κατά Συγχαρητήρια στην κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και eh, ε, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, μια πρόταση για την τροποποίηση της πράξης 20 Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Η κυρία Γκομάη είναι συγγήτρια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Τόμσον. Παρακαλώ κυρία Τόμσον, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρους της κυρίας Γκόμαϊ να διαβάσω τα δικά της σχόλια πριν από την ψηφοφορία. Είναι υπεύθυνη για το gender mainstreaming στην Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων και θα ήθελα να ζητήσει την υποστήριξη της έκθεσης όσον αφορά την τροποποίηση του νόμου που αφορά ε, της πράξης ε, ε, που αφορά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία προκειμένου να ενισχυθούν οι πτυχές της ατζέντα προτείνει τις τροπολογίες ούτως ώστε να υπάρχουν ώστε να αποφευθεί να υπάρχουν πάνω από δύο υποψήφοι για την ίδια ατζέντα. Αυτή είναι η τροπολογία 1 και 3. Και στο κατάλογο αυτό για να υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών και υποψηφίων των εθνοτικών μειονοτήτων, θα ήθελε να προτείνει μια αναλογική εκπροσώπηση του φύλου και μια καλύτερη εκπροσώπηση των εθνοτικών μειονοτήτων και των υποψηφίων τους. Αυτή είναι η τροπολογία υπαριθμών 2. Ε, βουλευτές που είναι έγκυοι και πρόσφατα γέννησαν παιδιά ε, προσωρινά δεν θα πρέπει να αντικαθίστανται. Επίσης θα θέλει να διατυπώσει μια πρόταση ε, ούτω ώστε να αντικαθίστανται τα μέλη του Κοινοβουλίου σε περίπτωση, προσωρινά σε περίπτωση εγκυμοσύνης στο κετού ή υιοθεσία. Λοιπόν, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναβολή τη ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή, διότι από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποσυρθούν να αποσυρθεί η έκθεση διότι το βασικό θέμα δεν είναι η αντιπροσώπευση των φύλων στον κατάλογο αυτόν. Το θέμα ποιο είναι. Είτε συμφωνούμε με τον Ενωμένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο, τον ΙΕΟ, είτε όχι. δεν αποφασίστηκε κάτι ούτε στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Δεν ε, έχουμε θέμα για πολιτική συζήτηση κατά την άποψή μου πάνω σε αυτό. Ίσως είναι λίγο πρόημο να αποφασίσουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Γιανακουδάκη, να υποστηρίξω και εγώ αυτό το σχόλιο. Όταν το είδα το έγγραφο και ήρθε μπροστά μου, έξε πλάκιν. Δεν ήξερα ότι είχαμε συμφωνήσει να έχουμε έναν ευρωπαϊκό κατάλογο. Και αν δεν έχει κανεί κατάλογο, πώ μπορεί να έχει ποσοστώσει. Πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Εκτό αν η λίστα πέρασε, εγκρίθηκε χωρί να το προσέξω. Αλλά εξεπλάγει αρκετά. Καλύτερα λοιπόν να το αφήσουμε, το να βάλουμε για την ώρα. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ σκοπεύει στις 19 Νοεμβρίου να κάνει την ψηφοφορία. Είναι απόφαση των συντονιστών να υποβάλουμε δηλαδή τροπολογίες εμείς απευθείας στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Μπορούμε να ψηφίσουμε όμως ε, σχετικά με το αν πιστεύετε εσείς ότι πρέπει σήμερα να γίνει ψηφοφορία ή όχι. Αυτοί που επιθυμούν να ψηφίσουμε σήμερα, παρακαλώ να σηκώσουν τα χέρια τους. Αυτοί που πιστεύουν. Θα τα πω στα αγγλικά, λέει You Θέλετε να αναβάλλετε την ψηφοφορία εσείς και ε, νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία που επιθυμεί την αναβολή. Ωραία. Αποφασίσατε λοιπόν να αναβληθεί η ψηφοφορία. Okay. Εντάξει. Eh, Ωραία, περνάμε στο επόμενο τότε θέμα. Γυναίκες εργαζόμενες επισφαλής θέσης απασχόλησης. Έκθεση πρωτοβουλίας που αποφάσισαν οι συντονιστές. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα διότι ε, διάφορες οικονομικές ε, συνθήκες ε, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των επισφαλών θέσεων απασχόλησης για τις γυναίκες με κακή αμοιβή και ούτω καθεξής. Από πλευράς Επιτροπής μας η κυρία Τόμψεν είναι η συγγήτρια. Θα ήθελα να της δώσουμε το λόγο, παρακαλώ. Uh, Συμφωνώ μαζί σας Πολύ σημαντική είναι η έκθεση και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε. Θα αρχίσουμε λοιπόν. Uh, Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται Υπαλήθευση. για την 20 ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 20 The vote is closed. Πέρας. 20 έτσι. Εγκρίνεται 14 ψήφοι υπέρ 9 κατά. 21 υπέρ κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Όχι. Καλά, επαλήθευση. 21. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. The vote is closed. Πέρας. Ναι, εγκρίνεται. 19 προς 6. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, από την Επιτροπή Απασχόλησης 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έξι της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση σας παρακαλώ για την 24. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 προς 15. Η 4 της Επιτροπής Απασχόλησης. Α, καταπίπτει. Το ίδιο και 8. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση για την 31 υπέρ ε, συγγνώμη ψηφίστε So now ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 προς 13. 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ε, ε, η 1 της Επιτροπής Απασχόλησης την έχουμε ψηφίσει αυτήν, δεν την ψηφίζουμε μάλλον, ε, υπέρ, κατά, αποχές για την 30 για την 33 ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας. 13 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. Ε, η 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, επαλήθευση για την ε, συμβαστική 5. The Πέρας. Ναι, εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Ε, η τρία της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, 9 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 έτσι ίδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές Πρέπει να γίνει επαλήθευση. Για τη 41 παρακαλώ, ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρα. Απορρίπτεται 12 προς 13 ψήφοι. 42 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 ε, ε, της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, Συγγνώμη, Πρόεδρε. Εγώ έχω ψηφορεί στον προπολογισμό που ήταν πάρα πολύ μακρά με πολλέ ψηφορίε και πήγαινε πιο σιγά, πρόεδρο. Σε αυτή την επιτροπή που έχουμε λίγε ψηφοφορίε δεν καταλαβαίνω γιατί συστρέχεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ε, υπάρχει χρόνο. Δεν έχουμε καν χρόνο να γυρίσουμε τη σελίδα και να καταλάβουμε. Ακούω και του διερμηνίε που μιλάνε γρήγορα. Ε, λίγο ηρεμία, κυρία Πρόεδρε. Τι να σα πω δηλαδή. Υπάρχει διαφορά μεταξύ προπολογισμού και επιτροπή γυναικών. Όπου ο πρόεδρο. Ε, εκεί είχαμε σωρό ολόκληρο τροπολογιών και στην άλλη επιτροπή μιλάει αργά ο πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτά είχα να πω. Okay. I will try to... Ε, Καλά. Θα προσπαθήσω να μιλάω πιο αργά. Αλλά ε, θα ήθελα όντω να μου λέτε ε, πώ επιθυμείτε να διεξάγετε η ψηφοφορία. Εγώ μπορώ να είμαι λίγο πιο αργή. Τώρα ακούστε με όλοι σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, παλήθευση. Ψηφίστε. 48 για 48. Ελπίζω όλοι να κατάλαβαν ότι ψηφίζουμε για την τροπολογία 48 πέρα της ψηφοφορίας 26 ε, ψήφοι υπέρ εγκρίνεται λοιπόν και τώρα φίλοι μου να συνεχίσουμε την ψηφοφορία για την 49 τώρα θα ψηφίσουμε παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα αν συμφωνείτε, ας περάσουμε συμβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση για την τροπολογία 5. Παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. πού And uh, it's rejected. Απορρίπτεται 12 υπέρ, 14 κατά. Συνεχίζουμε. Θα έρθουμε λοιπόν στην τροπολογία της Επιτροπής Απασχόλησης Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Ε, β από την επασχόληση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε τον υπαριθμό 10 υπέρ κατά αποχές θα γίνει επαλήθευση για τη 10 άρχεται η ψηφοφορία The τη ψηφοφορία. της ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 ψήφοι κατά και 12 ψήφοι υπέρ 11 υπαριθμών 11 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε. κατά αποχές εγκρίνεται F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 12 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει επαλήθευση υπέρ άρχεται η ψηφοφορία για την 12 πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 18 ψήφι υπέρ 8 κατά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 με 21 ψήφους υπέρ και 4 ψήφους κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, την κυρία Τόμσον. Τόμσεν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών. Προχωρούμε τώρα ε, στο σημείο 10 της μέσης διάταξης. Τίτλος ε, «Συμβολή των πολιτικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων. Θα γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Ζαμπόρσκα. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας στις 24 ε, ε, Νοεμβρίου το αποφάσισαν οι συντονιστές. Έχουμε και έγγραφο εργασίας που έχει μας έχει παρουσιάσει η συγγητριά μας. Έχουμε κάνει και μια πρώτη συζήτηση. Στις 23 Ιουνίου ήρθαν ε, και εμπειρογνώμονες. Επίσης μιλήσαμε για την αγωνική ε, ευθύνη και την επένδυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για να, ε, προληπτικούς λόγους, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων. Η συγγήτριά μας, κυρία Ζαμπόσκα, θα πάρει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την, ε, παρουσία, την εισαγωγή στην έκθεσή μου σε σχέση ε, με τη συμβολή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση εγκληματικότητα των νέων. Ήδη ευθύ εξ αρχής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις ε, εισφορές σας, τις συμβολές κατά τη διάρκεια της ε, πεφορικής ακρόασης που είχαμε διοργανώσει πρόσφατα. Οι συμβολές αυτές ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες και προσπάθησα πραγματικά να συμπεριλάβω ορισμένες από αυτές στην έκθεσή μου η διεύθυνση εξ αρχής θα ήθελα να σημειώσω ότι το θέμα αυτό είναι επίμαχο κάτω από μια ορισμένη άποψη και αυτό φάνηκε καθαρά και στην ακρόαση γιατί εκεί ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις εν σχέση με το πώς η οικογένεια μελλοντικά μπορεί να επηρεάσει τους νέους και πώς επίσης επηρεάζει και διαμορφώνει την ε, νεανική εγκληματικότητα. Το είπα και θα ήθελα να το επαναλάβω. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε κάποιες παρανοήσεις, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως έκανα στην έκθεσή μας, τα διεθνή ε, πολιτικά και θεσμικά όργανα όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΠΟΕ. η Παγκόσμια Συγγνώμη Οργάνωση Υγείας, ούτως ώστε να αποφευθούν ε, τυχόν ε, παρανοήσεις. Ε, στο θέμα αυτό αφιερώνεται η διεθνής ε, προσοχή, η παγκόσμια προσοχή, γιατί υπάρχει μια αύξηση στην εγκληματικότητα των νέων και υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι που διαπράττουν ε, εγκληματικές πράξεις από τη μία. Από την άλλη, η εγκληματικότητα περιλαμβάνει νέους όλο και μικρότερης ηλικίας και υπάρχει και μία αύξηση της βίας. Ενώ οι διαστάσεις της ε, βίας μεταξύ των νέων είναι παρόμοιες με αυτές που παρατηρούμε στους ενηλίκους. Συχνά τονίζεται η ευθύνη των, της οικογένειας, των γονέων συγκεκριμένα, αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος του παιδιού, και φυσικά ο περίγυρος παίζει ένα ρόλο. Και σε αυτό συνηγορούν και τα συμπεράσματα εκθέσεων διακεκριμένων ε, διεθνών οργανισμών. Ωστόσο, δίδεται και κάποια προσοχή στο πώς η οικογένεια, στο πώς κατοχυρώνεται η οικογένεια, η οικονομική βάση, πώς διαμορφώνεται η οικονομική βάση της οικογένειας, ούτως ώστε τα παιδιά να διαβιούν σε ένα υγιές περιβάλλον. Γιατί τα παιδιά αυτά, εάν μεγαλώσουν σωστά, τότε είναι εξασφαλμένο το μέλλον τους για την κοινωνία. Ε, δίδεται λοιπόν λίγη προσοχή στο πώς εξασφαλίζουν οι γονείς τις προϋποθέσεις για να μεγαλώσει το παιδί σε ένα υγιές περιβάλλον. Ε, προκειμένου να τονιστεί περισσότερο αυτή η πτυχή, ε, τονίζω τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και το, της ίσης των φύλων, ε, καθώς και της επίτευξης μιας ισορροπίας μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Επίσης θα ήθελα να σε ψήσω την προσοχή στο γεγονός ότι στον τομέα αυτό ότι το τομέας αυτό συχνά παραμελείται, δεν του δίδεται αρκετή προσοχή. Σύντομα θα συζητήσουμε και το θέμα των κινδύνων από το ίντερνετ για μια υγιή εξέλιξη των νέων επίσης για ζητήματα σεξουαλικής κατοικοποίησης και εκμετάλλευσης μικρών παιδιών. Σε σχέση με την επόμενη έκθεση συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και εδώ βλέπουμε ότι τα φαινόμενα αυτά αυξάνονται όλο και περισσότερο. Χθες ε, ακούσαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης πώς ασκείται η βία κατά των παιδιών, όχι μόνο εκ μέρους ενηλίκων, αλλά και πολύ συχνά είναι τα ίδια τα παιδιά δράστες άσκησης σεξουαλικής ε, βίας και συνεπώς ε, διαπράττουν τα ίδια τα παιδιά εγκληματικές ε, πράξεις. Στην έκθεσή μου ήθελα επίσης να σας επισημάνω το γεγονός ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να λάβουν τη δική τους ευθύνη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα συγκεντρωτισμό της πολιτική ευθύνη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά. Θα πρέπει και οι κράτες, τα κράτη-μέλη να λάβουν τις ευθύνες τους. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατόν να συντονίσει, να υποστηρίξει μάλλον τις επιμέρους πρωτοβουλίες των χωρών μελών μέσω οικονομικής στήριξης διαφόρων προγραμμάτων τα οποία επιλέγουν ή εκπονούν οι διάφορες κυβερνήσεις ή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τον τομέα των γονεϊκών ευθυνών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η οικογένεια είναι η πιο, ο πιο σημαντικός παράγων για την ανατροφή των παιδιών, χωρίς να είναι η μοναδική επίδραση και συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν είναι η πιο καθοριστική επίδραση αυτή των γονέων. Γι' αυτό αναφέρω στην έκθεσή μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παίζει σημαντικό ρόλο τονίζοντας ακριβώς ε, και χαρά στις πολιτικές ή μεταχειρήσεις των φίλων. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για τα παιδιά αλλά και για άλλα πρόσωπα τα οποία ε, τα φροντίζουν. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε σε μια πλατύτερη βάση, σε ένα πλατύτερο κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο γιατί αυτό είναι το περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Τελευταία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ορισμένες εκθέσεις ε, που ε, τονίζουν τη δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη η οποία θα πρέπει να λεφθεί σοβαρά υπόψη όχι μόνο λόγω της γύρανσης του πληθυσμού αλλά και λόγω του γεγονότος ότι έρχονται όλο και λιγότερα παιδιά στον κόσμο. Δηλαδή, τα μικρά παιδιά πλέον είναι κάτι το πολύτιμο. Επειδή ακριβώς ε, τα παιδιά αυτά θα εξασφαλίσουν την οικονομική ε, εξέλιξη Γι' αυτό δεν μπορεί να μας είναι αδιάφορος ο περίγυρος εντός του οποίου μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά, τα οποία θα εξασφαλίσουν τη μελλοντική κοινωνία. Πρόκειται για παιδιά τα οποία υποπέπτουν σε εγκληματικές πράξεις. Και εφόσον συμβαίνει αυτό, τα παιδιά αυτά ε, θα συνιστούν ένα οικονομικό έλλειμμα για την κοινωνία γιατί δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν κανονικά σε αυτήν και θα παραμείνουν ένα βάρος για την κοινωνία, ένα φορτίο. Αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει να σχηματίσουμε την εντύπωση ότι ο περίγυρος της περισσότερης οικογένειας είναι αρνητικός, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι νέοι ε, μεγαλώνουν αρμονικά σε υγιείς οικογένειες και θα συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση της ε, μελλοντικής κοινωνίας. Θα ήθελα παρόλα αυτά να σε επισημάνω ότι πράγματι αυξάνεται η εγκληματικότητα των νέων και συνιστά όλο και περισσότερο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι προσπάθησα στο πλαίσιο της έκθεσής μου δεν ακούμε πλέον την ομιλήτρια, έχει κλείσει δυστυχώς το μικρόφωνο της φαίνεται. Προσπάθησα λοιπόν ούτω ώστε να απευθύνει μια σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τις χώρες μέλη. Ούτως ώστε να εξεταστεί η εισφορά, η συμβολή των ε, γονέων από οικονομική άποψη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αναθέσει κάποιες έρευνες διεξογειορισμένων μελετών που να ασχολούνται σαφώς με αυτό το τομέα. Δηλαδή, τι σημαίνει από οικονομική άποψη όταν μια οικογένεια μπορεί να εξοπλίσει σωστά το παιδί, ο νέος δεν διαπράβεται εγκληματικές πράξεις και αντίθετα εντάσσεται σωστά στην κοινωνία. Πώς όλα αυτά αντανακλώνται σε αριθμούς τι σημαίνει διαμόρφωση ενός θετικού περιβάλλοντος σε αντίθεση με τη διαμόρφωση ενός αρνητικού για τα παιδιά περιβάλλον ε, τα οποία στη συνέχεια θα γίνουν ε, εγκληματίες ή θα παραβατικοί. Ε, και θα επανέλθω στην αρχική μου φράση. Όταν απαιτούμε από τους γονείς να αναλάβουν τα γονικά τους καθήκοντα, θα πρέπει από την άλλη να δούμε να σκεφτούμε ότι είναι στη θέση να εξασφαλίσουν και τα, να ασκήσουν τα γονεϊκά τους δικαιώματα, δηλαδή είναι οικονομικά ανεξάρτητοι. και δεν επηρεάζονται από ορισμένους αρνητικούς παράγοντες που ενδεχομένω θα είχαν αρνητική επίδραση στα παιδιά τους. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεσή μου και θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν με παρατηρήσεις και τις δικέ τους ιδέες στον εμπλουτισμό της έκθεσής μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Ζαμπόσκα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση είναι η κυρία Κώστα στον κατάλογο. το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Άννα Ζαμπόρσκα, για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση που έχει πολλές πτυχές και πολλές σημαντικές αναφορές. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ανησυχία της και την μέρημνά της να αποκτήσει μεγαλύτερη ευθύνη η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις συνθήκες τις συγκεκριμένες που μπορούν να δημιουργηθούν ούτως ώστε ο χρόνος εργασίας και ο οικογενειακός χρόνος και δραστηριότητα των ανδρών και των γυναικών μπορούν ε, να συμφιλειωθούν καλύτερα και να μπορούν να ασκήσουν τα γονικά τους καθήκοντα οι άνθρωποι περισσότερο. Ε, διότι πολύ συχνά περιορίζονται πολύ και σε χώρο και σε χρόνο οι γονείς. Αυτό θέτει το σημαντικό θέμα της αναγνωρίσεως, της αξίας της δουλειάς της μέρημνας, της φροντίδας και στη διάσκεψη του Πεκίνου και σε άλλα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών υπενθυμίζω ότι ζητήθηκε να υπάρχει στο ΑΕΠ δίπλα στους οικονομικούς δείκτες τους κλασικούς που ζητάει και Άννα Ζαμπόρσκα να υπάρχει και μια αξιολόγηση και οικονομικής φύσεως της αόρατης δουλειάς που είναι μια μεγάλη πηγή ε, κοινωνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς η πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων να συνδεθεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα από πλευράς ε, των γονέων. Αυτό που θα μπορούσα να προτείνω είναι μεγαλύτερη προσοχή σε άλλες πηγές που θα μπορούσαν να ε, στην υποστήριξη των οργανώσεων για τους νέους. Δίπλα στην οικογένεια, πέρα από την οικογένεια υπάρχουν και άλλοι φορείς εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν περισσότερα και μπορούν να καλύψουν ένα κενό, το κενό χρόνο που έχουν τα παιδιά καμιά φορά και οι νέοι, ε, υποστήριξη ε, αυτών των φορέων που μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά πέρα από τους γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε τους όρους του Eurostat όσον αφορά την εξέταση αυτών των συνεισφορών στο ΑΕΠ και θα πρέπει να δούμε πόσο κοστίζει στην κοινωνία η έλλειψη της παρουσίας της πολιτισμικής αν θέλετε και πόσες δυσκολίες και πόσο κοστίζουν οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε, όπω είναι οι μονογονικέ οικογένειε, που οι γυναίκε είναι οι μόνοι γονεί και χρειάζονται υποστήριξη. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, όπω είπατε, όσον αφορά τα ωράρια, όσον αφορά το να βοηθήσουμε αυτέ τι μητέρε. Ζητούν οι γυναίκε ευελιξία. Και τελικά η απάντηση ήταν η προσωρινή εργασία. Δεν θέλαμε αυτή την ευελιξία. Θέλαμε ευελιξία των ωραρίων και τη οργάνωση τη εργασία που να ταιριάζει με τι οικογενειακέ υποχρεώσει να νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα ποιες άλλες συνθήκες μπορούν να υπάρξουν που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων κοινωνικών. Δεν μπορούν να είναι όλες τι πλάτες της οικογένειας, που σήμερα οι πλάτε είναι πια στην Ευρώπη, οι πλάτη της οικογένειας. Χρειάζεται μεγαλύτερη αντιμετώπιση και το θέμα των εξαρτήσεων. Εξαρτήσεως των νέων από το αλκοόλ, από το ναρκωτικό, από τη μείωση της προσοχής της γενικής που δίδεται όσον αφορά τους τρόπους ζωής. Και αυτά δημιουργούνται πολλές φορές από την αγορά αυτές τις συνθήκες. Μειώνεται η προσοχή στα κράτη-μέλη όσον αφορά τον αλκοολισμό των νέων, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και την κοκαίνη. Χρειάζεται πιο ολοκληρωμένη πολιτική που θα πρέπει να θετηθεί προς πιο σοβαρές κατευθύνσεις και μέτρα. Και με την ε, ανασφάλεια στην εργασία υπάρχει, και αυτό είναι ένα ως δημιουργεί πρόβλημα. Και η εγκατάλειψη, υπάρχει η διασύνδεση μεταξύ της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου από πλευράς τους νέους με την αύξηση της εγκληματικότητας των νέων. Πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσφορά από τα κράτη-μέλη αυτό το προβλέπει άλλωστε και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ε, κατάρτιση. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να υποστηριχθεί η οικογένεια σε αυτό, δηλαδή να μειωθεί η πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου από τα παιδιά. Αυτό είναι τα στοιχεία που επηρεάζει την αύξηση της εγκληματικότητας των νέων. Συμφωνώ να δημιουργηθεί ένα δίκτυο προστασίας και βοήθειας για τις οικογένειες, σωστό αυτό, και πρέπει να αξιολογήσουμε και τι συνέπειες έχουν οι πολιτικές ετρικογενειών. Δεν είμαι αντίθετη. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης. Μεταγενέστερη υποστήριξης. Πολύ συχνά οι οικογένειε είναι εύθραυστε, είναι μονογονικές, αντιμετωπίζουν δυσκολίε Εντός τους να έχουν πραγματική αυτονομία και πραγματικές δυνατότητες. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για την παιδεία και για τι ενώσει των νέων και για πολιτικές που θα μειώνουν και θα προλαμβάνουν τις διάφορες εξαρτήσεις από διάφορα πράγματα που έχουν αυξηθεί πολύ μεταξύ των νέων. Παραδείγματα στην Ιταλία, κατά την άποψή μου, τα τελευταία χρόνια ζητείται να γίνουν πολλά περισσότερα για να μειωθεί ο αλκοολισμός των νέων και να προληφθεί. Έχουμε φοβερά στοιχεία στη χώρα μας. Οι, οι νέοι κάτω από 13 είναι οι μεγαλύτεροι πότες της Ευρώπης. Εμεί δεν είχαμε πριν από 10 χρόνια τέτοιο πρόβλημα αλκοολισμού. Δεν δόθηκε η προσοχή τα τελευταία χρόνια στον τομέα και πλευρά των κυβερνήσεων και αυτό φταίει. Θα πρέπει ζητήσουμε από του θεσμού να επιληφθούν του θέματο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σιμίσκιν τώρα και μετά η Σοφή Ιντβέλτε. Η κυρία Σινέσκιν. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, πρέπει να φύγω ευθύ αμέσω μετά την παρέμβασή μου. Δεν είναι πάρα πολύ ευγενικό αυτό, αλλά μακρηγόρησαν οι συνάδελφοι. Δυστυχώ στην προηγούμενη συζήτηση δεν ήμουν παρούσα, γιατί αλλιώ ε, θα είχα αναρωτηθεί αν ε, ευστοχεί η σύνταξη τη έκθεση η ίδια. Δηλαδή, ε, περί τίνο ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποια πράγματα δεν έχει καμία ευθύνη. Δεν καταλαβαίνω καν τη θέση του ΕΛΚ. Αν δω όλο τον κατάλογο των ζητημάτων ε, που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα αφενό ε, και με τα οικογενειακά ζητήματα αφετέρου, που προσπαθήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο να πραγματευτούμε. Ε, λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει ασυνέπεια στη θέση τη ομάδα. Το ΕΛΚ, παραδείγματο χάρη, ισχυρίζεται ότι οι οικογένειε όσων έχουν αλλάξει φύλλο δεν είναι θέμα αρμοδιότητα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάκριση στο θέμα του γάμου αυτών των ανθρώπων, η μονογονιακή εθνικές οικογένειες, η ελευθερία των θρησκευτικών πεπιθήσεων, διασυνοριακά δικαιώματα ω προ το διαζύγιο, ε, μαζικά σκάνδαλα κακοποίηση παιδιών, διεθνεί και καλυμμένε επιχειρήσει. Όλα αυτά δεν τα συζητάμε εδώ, αλλά συζητάμε πώ θα μεγαλώσουν τα παιδιά του οι γονεί, αν υπάρχει κάτι που είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων, είναι ακριβώ αυτό, πώ θα αναθρέψουν τα παιδιά του και συγγνώμη, αλλά ε, διαβάζοντας την έκθεση για μένα προσωπικά λέει μέσα effective parenting, ε, ε, ε, αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του γονέα. Μα συγγνώμη, αυτό είναι θέμα ηθικής. Όλοι δικαιούνται να έχουν την άποψή τους. Αλλά εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε καμία δουλειά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσουμε τι εστί αποτελεσματικός γονιός. Όλοι θα αποφασίσουν πώς θα αναθρέψουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν δύο-τρεις παράγοντες παράγραφοι μέσα στην έκθεση, πρόεδροι, συγγνώμη, αλλά καταδεικνύουν ένα φόβο ενώπιον τη σύγχρονη εποχή. Ε, κατά τη γνώμη μου, ε, ε, έχουμε πλησιάσει οριακά στην ιστερία. Ε, πάντοτε υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και πάντοτε θα υπάρχουν. Σήμερα δεν υπάρχουν περισσότερε απειλέ σε σχέση με το παρελθόν ή σε σχέση με το μέλλον. Α είμαστε λοιπόν ρεαλιστέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μπει στα χωράφια των γονέων εκείνοι θα αποφασίσουν πώ θα αναθρέψουν τα παιδιά του. Σας ευχαριστούμε κυρία Σοφή Ιντβέλτε. Η κυρία Σένσιν ε, τώρα. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. E, ναι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση διάβασα πολλές ενδιαφέρουσες συστάσεις σε αυτή την έκθεση. Ωστόσο, πολλές ε, πτυχές που ανήκουν στο θέμα αυτό δεν έχουν ληφθεί υπόψη ή δεν παρουσιάζονται με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Από, τις, από τα όσα υπόθηκαν σήμερα προκύπτει ότι η συγκήτρια έχει συγκεντρωθεί μόνο στο ρόλο της οικογένειας όσον αφορά την πρόληψη της εγκληματικότητα. Και αν η έκθεση έφερε αυτόν τον τίτλο, ίσως οι παρατηρήσεις μου θα ήταν άστοχες. Αλλά η έκθεση φέρει έναν διαφορετικό τίτλο, που είναι η συμβολή των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης έτσι λοιπόν θα πρέπει να διερωτηθούμε ποια μπορεί να είναι η δική μας ε, συμβολή και ε, εάν ε, είναι ανεπαρκής θα πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί. Πράγματι χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική πολιτική για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Χρειαζόμαστε την οικογένεια καθώς και το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο καθώς και την εκπαίδευση η οποία συμβάλλει εδώ, προωθεί κάτι τέτοιο, καθώς... Ε, αλλά η συγκίτρια, συγγνώμη, ε, συγκεντρώνεται στην ευθύνη των γονέων. Νομίζω ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος της εκπαίδευσης, του σχολείου, των οργανώσεων νέων, που επίσης ε, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων. Η γονεϊκή υποπτία δεν είναι αρκετή για να προστατεύσει τους νέους από την εγκληματικότητα. Οι νέοι κατατείνουν προς την αυτονομία, την ανεξαρτησία κλπ. Και αυτό είναι εντελώς αυτονόητο. Ακόμα και οι γονείς που έχουν πλήρη συνείδηση των ευθυνών τους δεν μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν εδώ την οικογένεια αλλά και το σχολείο καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικέ προποθέσει και επιτρέψατε μου να σα αναφέρω ένα παράδειγμα από τον τομέα του αθλητισμού. Έχουμε πολύ καλές εμπειρίες με το box. Κάποιος προπονητής ε, διάλεξε παραβατικούς νέους, τους μάζεψε από το δρόμο και τους ε, πρότεινε αντί να δέρνονται στο δρόμο να εξασκηθούν στο box η ίση, ο τομέας της ίσης μεταχείρισης για την, των φίλων για την ε, καταπολέμηση του νεανικής εγκληματικότητας δεν μπορεί να περιοριστεί ε, στο ζήτημα της γονεϊκής ευθύνης. Αλλά εξαρτάται επίσης από την εξασφάλιση κάποιων γνώσεων όσον αφορά την ίση μεταχείριση των δύο φίλων, Δηλαδή πρέπει να αποφευθούν μέσω της εκπαίδευσης οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα καθώς και ο ρόλος των φίλων. Θα πρέπει να προωθηθεί η δυνατότητα ενσυναίσθησης των, ε, μεταξύ των νέων και στο σχολείο. Εάν θέλουμε να αναπτύξουμε κάποιες δεξιότητες τους νέους και μια μεγαλύτερη συνειδητότητα, θεωρώ ότι αυτό θα συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της ε, εγκληματικότητας των νέων. Θα πρέπει να εκπονήσουμε κάποια προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτών είναι δυνατόν να διαμορφωθεί σωστά η προσωπικότητα, το αυτοαίσθημα και ο σεβασμός των άλλων στους νέους και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται ζητήματα φύλου στην ε, ε, παιδαγωγική τους. Τα στατιστικά στοιχεία μας λέει ότι σε μεγάλο βαθμό νέοι εγκληματίες είναι ανεπιθύμητα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε λεγόμενες ψυχρές ε, οικογένειες, σε ψυχρές συνθήκες. Αποστρέφονται τον κόσμο και έτσι το έγκλημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φυσική συνέπεια της κατάστασής τους. Πολύ συχνά είναι οι ίδιοι θύματα ε, γονεϊκής βίας ή γονεϊκής παιδοφιλίας. Πολύ συχνά οι γυναίκες εκτίθενται σε μορφές βίας εντός της οικογένειας και αυτό αφορά και νέους και παιδιά. Ε, παιδιά και νέοι θα πρέπει εν μέρη να προστατεύονται από τους ίδιους τους γονείς και από την ίδια τους την οικογένεια. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής θα πρέπει οι νέοι να έχουν μια καλή πρόσβαση στις γνώσεις, στις θέσιμες γνώσεις για τη σεξουαλικότητα, για σύγχρονα για σύγχρονες ε, ε, ε, πρόληψης, προφύλαξης κλπ. Υπάρχουν... Ε, θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του κόστους που θα πρέπει να καλύψει η κοινωνία σχέση ακριβώς με μορφές νεανικής εγκληματικότητας. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στην ε, ελληπή γονεϊκή ευθύνη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να οροθετηθεί η γονεϊκή ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Και διαρωτώ με τι γίνεται σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τι στοιχεία έχουμε εδώ εν σχέση με την επίδραση που ασκούν οι γονείς σε συνάρτηση με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων. Ε, ίσως η εισηγήτρια θα πρέπει να διευκρινίσει καλύτερα αυτό το τμήμα της εισήγησης, της έκθεσής της. Πράγματι ισχύει ότι η βελτίωση των οικονομικών ε, συνθήκων ε, αυξάνει την συνειδητοποίηση των γονέων παρόλο που η σχέση αυτή δεν είναι πάντοτε σήμαντη. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με την καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας σε συνάρτηση με τα φύλλα. Επίσης δεν έχουμε πληροφορίες σε σχέση με τις εμπειρίες των δύο φύλων στο πλαίσιο της εγκληματικότητας των νέων. Είναι απολύτως δυνατό κάποια ορισμένες μορφές της εγκληματικότητας να διαπράττονται από γυναίκες ή από νέες και άλλες μορφές εγκληματικότητας από νέους. Και συμμερίζομαι την άποψη της εισηγήτρια ότι θα πρέπει να έχουμε στοιχεία και από τις οργανώσεις των νέων. Εγώ θα καταθέσω τις δικές μου τροπολογίες και τις δικές μου παρατηρήσεις. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε επικεντρωθεί